So, ladies and gentlemen, dear colleagues. Συνάδελφοι, νομίζω πως θα πρέπει να ξεκινήσουμε. Ονομάζομαι Πέτα Λίζα και μου ζητήθηκε ήδη από τους ε, συναδέλφους καθόμενες είμαι το παλαιότερο μέλος της Επιτροπής. Ελπίζω να μην είμαι βέβαια, αλλά μου το είπαν ότι είμαι το παλαιότερο μέλος της Επιτροπής ΕΝΒΗ και καθώς δεν αποτελούν πλένη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ο πρώην πρόεδρος και αντιπρόεδρος και επειδή άλλος συνάδελφος ε, του Προεδρίου ε, συμμετέχει πλέον στην Ήτρε, μου ζητήθηκε από εμένα να προεδρεύσω προσωρινά σε αυτή τη συνεδρίαση. Έχω εδώ μπροστά μου τις ε, σημειώσεις μου στα γερμανικά, στη γερμανική γλώσσα. Επειδή πρόκειται για ένα τεχνικό και ε, νομικό ζήτημα, οπότε αν δεν καταλαβαίνετε τη γερμανική γλώσσα θα ήθελα να φορέσετε τα ακουστικά σας. Ε, Κυρίσω λοιπόν την έναρξη της συνεδρίασής μας ε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Ο στόχος της σημερινής συνεδρίασης είναι να εκλέξουμε τον πρόεδρο της Επιτροπής Περιβάλλοντος Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων και να εκλέξουμε του τέσσερι αναπληρωτέ προεδρού. Καταρχήν θα πρέπει να διευκρινίσουμε το ποιο έχει το δικαίωμα ψήφου σήμερα εδώ. Φυσικά είναι τα τακτικά μέλη που έχουν εκλεγεί, σαφέστατα. Και έχουμε τέσσερις συναδελφούς που είναι τακτικά μέλη, αλλά δεν είχαν τη δυνατότητα να περιβρεθούν σήμερα εδώ και έχουν ορίσει αναπληρωματικούς. Οπότε η ΑΕ μας έχει πει, αντί για τον η κυρία Ολυρία Μιλέ θα πάρει το λόγο για λογαριασμό του ή θα ψηφίσει για λογαριασμό του Ανδρέας Λουκ. Το ECR μας είπε ότι για λογαριασμό ε, του κυρίου Ρομπ Ρούκεν η κυρία Ντέις Μελμπέρντ θα πάρει το λόγο και θα ψηφίσει και από τους μη εγγεγραμμένους δύο αλλαγές έχουμε εδώ για λογαριασμό του James Alexander Λέξη, ο Πιέρο Νίκολα Πεντιτσίνη θα ψηφίσει και επίσης για λογαριασμό της Κριστίλα Τσέλα ο κύριος Πουκ θα ψηφίσει. Υπάρχουν άλλα τακτικά μέλη τα οποία δεν είχαν τη δυνατότητα να παρευρεθούν στη σημερινή συνεδρίαση και όρισαν κάποιον για να τους εκπροσωπήσει. Δεν βλέπω να υπάρχει κανείς. Θεωρούμε λοιπόν πως ε, έχουμε εδώ αυτό το δικαίωμα ε, ψήφου για τακτικά μέλη και τους τέσσερις εκπροσώπους. Τώρα, για να έχουμε απαρτία πρέπει να διαπιστώσω ότι έχουμε απαρτία, δηλαδή το 1 τέταρτο των μελών, που σημαίνει 19 μέλη και βλέποντας εδώ την αίθουσα διαπιστώνω ότι έχουμε απαρτία. Οπότε θα ήθελα να ρωτήσω αν έχουμε υποψηφίους για την Προεδρία. Και για να οριστεί μια υποψηφιότητα θα πρέπει να υποστηρίζεται είτε από μια πολιτική ομάδα είτε από το 1 20 των μελών, δηλαδή 4 ε, μέλη τουλάχιστον. Νίλ Στόρβαλντ έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε για να είμαι σίγουρος ότι θα με αντιληφθείτε θα προσπαθήσω να μιλήσω στα γερμανικά. Και γιατί τα αγγλικά με δυσκολεύουν. Για την ε, πολιτική ομάδα New Europe προτείνω τον Πασκάλ Καφέ. Καλώς. Καθώς ε, τον ορίζετε ως υποψήφιο εκ μέρους της δικής σας πολιτικής ομάδας. Ε, δεν υπάρχει πρόβλημα. Ρωτώ λοιπόν ε, τον υποψήφιο αν πράγματι αποδέχεται την υποψηφιότητα. Καταφατικό νεύμα. Καλώς. Η κυρία Μύρια Μντάρη τώρα εκ μέρους των σοσιαλιστών ζητάει το λόγο. Παρακαλώ. Ναι. Πρωτού ε, περάσουμε στην πληροφορία. να αναφερθώ σε αυτό που είπατε για τους εκπροσώπους των τακτικών μελών. Η Μαρία Ρένα λοιπόν ε, θα αντικαταστήσει τη Ροβάνα Πλάν γιατί δεν έχει ε, φέρει σήμερα μαζί της την κάρτα για την ψηφοφορία. Οπότε ε, θα ήθελα να σας παρακαλέσω να λάβετε υπόψη σας λοιπόν αυτή την αντικατάσταση. Καλώς λέει ο Πρόεδρος, το λαμβάνουμε υπόψη μας και συνεχίζω τώρα στα γερμανικά και πάλι. Άρα λοιπόν ο υποψήφιος είναι τακτικό μέλος της Επιτροπής, πληρείται αυτή η προϋπόθεση. Ρωτώ λοιπόν ε, κατά πόσο έχει υποβληθεί και η δήλωση ε, των οικονομικών συμφερόντων και σε ό,τι αφορά τον κώδικα διοντολογία. Ε, η γραμματεία με ενημερώνει ότι έχουν υποβληθεί αυτέ οι δηλώσει. Καλώ. Περνάμε λοιπόν τώρα στην ψηφοφορία. Ας κάνουμε μια δοκιμαστική ψηφοφορία για να είμαστε σίγουροι. Ε, να είμαστε σίγουροι ότι λειτουργεί λοιπόν καλά το σύστημα, να μην έχουμε κανένα πρόβλημα, να τα κάνουμε όπως το κάνουμε και στην Ολομέλεια. So, müssen eine Minute Περιμένουμε εδώ να εμφανιστεί στην οθόνη. So, put your card into the machine. That's important. Βάλτε λοιπόν τις ε, κάρτες σας μέσα στο μηχάνημα, γιατί είναι σημαντικό αυτό. Αν δεν το κάνετε δεν μπορούμε να ξεκινήσουμε με την ψηφοφορία. <laughs> Okay, then Μπορούμε λοιπόν να περατώσουμε την ψηφοφορία. Τέλος λοιπόν της ψηφοφορίας. Δεν μπορώ να δω εδώ το αποτέλεσμα. Η γραμματεία μου λέει δεν υπάρχει πρόβλημα. Λειτουργήσε καλά το σύστημα. Την επόμενη φορά θα επαγρυπνώ περισσότερο. Αλλά εντάξει, δοκιμαστική ήταν η ψηφοφορία. Λοιπόν, τώρα θα πρέπει να αποφασίσουμε ως προς τον τρόπο της ψηφοφορίας. Εάν τουλάχιστον το 1 πέμπτο των μελών ε, επιθυμεί να γίνει μυστική ψηφοφορία, τότε θα το κάνουμε. Σε διαφορετική περίπτωση μπορούμε να ψηφίσουμε διαβοή. Οπότε ερωτώ, ε, υπάρχει κάποιο μέλος που να επιθυμεί μυστική ψηφοφορία. Δεν βλέπω να ζητάει κανεί το λόγο, οπότε για την υποψηφιότητα του κυρίου Πασκάλ Καφά. Διαβοή. Σας ευχαριστώ πολύ. Ε, τα θεμά μου συγχαρητήρια Πασκάλ για την εκλογή σας και νομίζω πως μπορείτε να αναλάβετε τα καθήκοντά σας. Οπότε εγώ επιστρέφω στη θέση μου ως μέλος της Επιτροπής και Πασκάλ πώς να συνεχίσει ως πρόεδρος. Well, thank you very much for... Ευχαριστώ πολύ που με εμπιστευτήκατε να προεδρεύω της Επιτροπής αυτής. Θα πω δύο λόγια, ξέρω ότι πιέζει ο χρόνος. Το πρώτο μήνυμα που θέλω να σας μεταφέρω είναι ότι η Επιτροπή αυτή τώρα είναι η μεγαλύτερη Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για πρώτη φορά. Και βέβαια αυτό είναι συμβολικό, όμως, όπως ξέρετε, στην πολιτική και τα σύμβολα έχουν σημασία. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι πρόκειται για ένα σύμβολο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που τι λέει, λέει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παίρνει πάρα πολύ στα σοβαρά τα θέματα του κλίματος, του περιβάλλοντος, των καταναλωτών, αν μη τι άλλο πολύ περισσότερο από ό,τι κατά το παρελθόν, όπως θα έπρεπε να κάνει και κανείς έχοντας υπόψη του πόσο πολύ επίγουν τα ζητήματα αυτά. Αυτό λοιπόν είναι ο πρώτος συμβολισμός και θα έπρεπε να κοινοποιηθεί σε όλα τα μέσα ενημέρωσης παντού ότι αυτή η Κοινοβουλευτική Επιτροπή είναι η μεγαλύτερη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για πρώτη φορά σε αυτή τη θητεία. Το δεύτερο μήνυμα που έχω να σας μεταφέρω είναι ότι θα είμαι πάρα πολύ προσεκτικός για το ότι δεν έχουμε μία Ανατολική και μία Δυτική Ευρώπη όταν μιλάμε για την μετάβαση. Στόχος μας είναι να προωθήσουμε την ουδετερότητα όσον αφορά το αποτύπωμα άνθρακα παντού. Μπορεί να ξεκινάμε από διαφορετικά σημεία κίνησης, αλλά πρέπει να φτάσουμε στο ίδιο σημείο, την ουδετερότητα όσον αφορά το αποτύπωμα άνθρακα. Και δεν πρέπει να μείνει καμία κατηγορία, καμία ομάδα, ε, κανείς πίσω. Αυτό λοιπόν πιστεύω ότι είναι ένα μήνυμα που πρέπει να μοιραστώ μαζί σας γιατί αποτελεί το DNA μας εδώ σε αυτή την Επιτροπή. Και το τελευταίο μου μήνυμα είναι ότι ε, θέλω να είμαστε στην πρώτη γραμμή, οι πρωτοπόροι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ε, στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, έτσι ώστε να διασφαλίσουμε ότι έχουμε το σωστό βαθμό φιλοδοξίας που δεν σημαίνει βέβαια ότι δεν θα γίνουν οι συμβιβασμοί, αλλά αν μη τι άλλο να είμαστε σίγουροι ότι ζητάμε αυτό που θέλουμε, αυτό που χρειαζόμαστε για να καταπολεμήσουμε την κλιματική αλλαγή, ε, να φροντίσουμε να προστατεύουμε το περιβάλλον κλπ. Όπου λοιπόν και αν κάθεστε σε αυτή την αίθουσα, σε όποια πολιτική ομάδα και αν ανήκετε, να ξέρουμε όλοι ότι μοιραζόμαστε το ίδιο μήνυμα. Και μην ξεχνάτε ότι οι νέοι έχουν το βλέμμα στραμμένο σε εμά και περιμένουν να δούνε τι θα κάνουμε. Σας ευχαριστώ. Αυτό λοιπόν ήταν το σύντομο μήνυμά μου ως εισαγωγή. Και τώρα ερχόμαστε στην επίσημη διαδικασία της ψηφοφορίας. Και τα είπε γερμανικά πριν ο Πέτερ το κομμάτι αυτό της διαδικασίας, θα το πω και εγώ στα γαλλικά, στη γλώσσα μου. Συνεχίζει στα γαλλικά λοιπόν ο κύριος Καλφά. Λοιπόν, περνάμε τώρα στην ψηφοφορία των αντιπροέδρων. Αρχίζουμε από την πρώτη αντιπροεδρία. Πρέπει να επαληθεύσουμε αν είναι οι ίδιοι αυτοί που ψηφίζουν. Υπάρχει κάποιος που άλλαξε, Μάργαρετ, υπάρχει κάποια αλλαγή. Δεν θα τα πω δανέζικα, και θα μπορούσα να τα πω δανέζικα, αλλά τέλος πάντων θέλω να συγχαρώ τον Καλφάν, αυτό θέλω να πω. Και χαιρόμαστε για την πρόθεση αυτής της συνεργασίας. Νομίζω ότι όλοι το θέλουμε αυτό, οι πράσινοι συμφωνούμε. Και Και προτείνω εδώ το συνάδελφο για την ε, πρώτη αντιπροεδρία. Και ξέρω ότι συμφωνεί. Μια στιγμή, περίμενε Μαργαρέτα, περίμενε, περίμενε, δεν φτάσαμε ακόμα εκεί. Έλεγα. Πρώτα απ' όλα, αυτοί που ψηφίζουν είναι οι ίδιοι, δεν υπάρχουν αλλαγέ. Ωραία. Επίση έχουμε πάλι απαρτία. Και τώρα ήρθε η στιγμή να ρωτήσω αν υπάρχουν υποψηφιότητε. Μάργαρετ. Συγγνώμη, συγγνώμη, βιάστηκα, δεν άκουγα πολύ προσεκτικά πριν. Συγγνώμη. Ένα σχόλιο έγινε εκτό μικροφώνου. Λοιπόν, συγχαρητήρια και πάλι και επαναλαμβάνω ότι προσβλέπουμε σε συνεργασία εδώ στην Επιτροπή αυτή. Οι προσδοκίες μας είναι μεγάλες να καταστήσετε το θέμα αυτό του περιβάλλοντος το πρώτο θέμα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ολόκληρο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Προτείνω λοιπόν τον Πασάχουλ ως πρώτο αντιπρόεδρο. Υπάρχουν άλλοι υποψήφοι? Όχι από ό,τι φαίνεται. Αν δεν ζητάει κανείς μυστική ψηφοφορία, τότε μπορούμε να ψηφίσουμε διαβοής για την πρώτη αντιπροεδρία. Ο Μπας του λοιπόν. Μπας, έλα εδώ. Λοιπόν, χωρίς εκπλήσεις, περνάμε στη δεύτερη αντιπροεδρία της Επιτροπής αυτής. Πάλι να δούμε αν παραμένουν οι, τα ίδια μέλη που ψηφίζουν. Δεν υπάρχει αλλαγή. Απαρτία έχουμε. Οπότε... Ρωτάμε τώρα τις πολιτικές ομάδες. Έχουν να προτείνουν υποψηφιότητες. Παρακαλώ. Ευχαριστώ και πρώτα απ' όλα συγχαρητήρια για τα νέα σας καθήκοντα και εμείς προσβλέπουμε σε συνεργασία μαζί σας. Εκ μέρους των σοσιαλιστών λοιπόν προτείνουμε τον Σεπ Ντάνστ στην δεύτερη αντιπροεδρία της Επιτροπής αυτής. Υπάρχουν άλλοι υποψήφοι? Ζητάει κανείς μυστική ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Όχι. Ωραία. Τότε μπορούμε να ψηφίσουμε, νομίζω, διαβοής για την δεύτερη αντιπροεδρία. Οπότε, καλό το Σεμπτάνς να έρθει εδώ μαζί μας. Πάμε τώρα σε θέση τρίτου αντιπροέδρου για την Επιτροπή. Ίδιος είναι ακόμα ο κατάλογος ψηφοφορίας, απαρτία. Έχουμε από τις ομάδες ο Πέτερ. Ευχαριστώ πολύ. Εν ονόματι του ΕΛΚ προτείνω Κρίστιαν Μπούζο, το συνάδελφο. Είναι έμπειρο μέλος της Επιτροπής αυτής είναι νομικός και γιατρός και έχει κάνει πολλά κατά το παρελθόν. Θα τον ψηφίσουμε αυτή τη θέση. Yeah. Άλλοι υποψήφοι. Από την πλευρά μου προτείνω είμαι νεοεκλεγένα τον Εύαν Μποσίνσιτς ήταν πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος στην Κροατία στο κρατικό κοινοβούλιο και τον προτείνω ως υποψήφιο για την θέση αυτή ε, του Αντιπρόεδρου. Ευχαριστώ. Άλλες υποψηφιότητες να ελέγξουμε σύμφωνα στους κανόνες, να ελέγξουμε αν τους υποστηρίζει η πολιτική ομάδα, τους υποψηφίους, αυτό ισχύει για το ΕΛΚ, ή από τουλάχιστον τέσσερα μέλη. Χρειαζόμαστε κατάλογο με τα ονόματα των τεσσάρων τακτικών μελών που ε, υποστηρίζουν τη δεύτερη υποψηφιότητα. Σηκώστε το χέρι σας παρακαλώ. Καλώς. Είσαστε πάνω από τέσσερις, είναι προφανώς αυτή η κατάσταση. Θα γίνει ηλεκτρονική ψηφοφορία για τη θέση τρίτου αντιπρόεδρου. Θα ξαναμιλήσω στα γαλλικά τώρα. Θα ξαναχρησιμοποιήσω τα γαλλικά. Πάρτε τις κάρτες σας παρακαλώ. Και ένα έτοιμα. Ξέχασα την κάρτα μου εκεί. Αν έχει την καλοσύνη να μου τη δώσετε παρακαλώ. Να η ελληνεγκή λοιπόν στην πράξη. Στην ομάδα Ρινιού. Ευχαριστώ πολύ. πρέπει να καθορίσουμε τα χρώματα για κάθε υποψήφιο. Με αλφαβητική σειρά. Ο κύριος Μπουζόη. Πράσινο κουμπί στα αριστερά. Και ο κύριος Σίντσιτς το κόκκινο κουμπί στα δεξιά. Ο κύριος Μπουζόη, πράσινος αριστερά, κύριος Σίντσιτς, κόκκινο δεξιά. Εντάξει. Μπορούμε να αρχίσουμε. Είναι όλα εντάξει. Ξεκινάμε λοιπόν την ψηφοφορία. Ψηφίστε παρακαλώ. Σας αφήνω μερικά δευτερόλεπτα να αλλάξετε γνώμη. Αν χρειάζεται ή να διορθώσετε κάποιο λάθος. 3, 2, 1, πέρας. Ο κ. Μπουζόη έλαβε 58 ψήφους, ο κ. Σίντσιτς έλαβε 15 ψήφους, σύνολο ψηφισάντων 74. Κύριε Μπουζόη, παρακαλώ να έρθετε εδώ. We are moving to the... Uh, Πάμε τώρα για την τελευταία ψηφοφορία για τον πέμπτο αντιπρόεδρο. Δεν υπάρχει ισορροπία όσον αφορά τα φύλλα, δεν υπάρχει πλήρη ισορροπία. Ξέρετε τον κανόνα. Έχουμε από το Ρινιού κάποιο αίτημα επίσημο. Πρόεδρε, απεχώρησε ένα μέλος μας, χρειαζόμαστε να πληρωτεί. Ο Ζαμπρόλ είναι εδώ και μπορεί να λειτουργήσει σε αυτή τη θέση αν συμφωνείτε. Καλώς. Τα τυπικά, καταρχήν. Για τον κατάλογο ψηφοφοριών, για τα μέλη, πέρα από την αλλαγή του ΡΙΝΙΟΥ τα άλλα είναι εντάξει. Οι ομάδες έχουν υποψηφιότητες για τη θέση του πέμπτου αντιπρόεδρου. Ορίστε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Συγχαρητήρια σε όλους τους εκλεγέντες. Θέλουμε διαφυλαχθεί ισορροπία των φίλων, να προτείνουμε ικανότατη αντιπρόεδρο, την κυρία Άνια Χάζενκαμπ, για θέση τέταρτης αντιπρόεδρου. Ευχαριστώ. Άλλες υποψηφιότητες υπάρχουν? Να υπενθυμίσω κάτι. Θα ξέρετε πιθανότατα ότι ο κανόνας είναι ότι χρειάζονται τουλάχιστον έναν άντα τέσσερις γυναίκες ή μια γυναίκα τέσσερις άντρες για την ισορροπία. Ευχαριστώ που δίνεται μια, προτείνεται μια γυναίκα, όχι να επιτευχθεί η ισορροπία των φίλων, δεν επιτυγχάνεται εδώ, αλλά τουλάχιστον να μην έχουμε κάτι που είναι τελείως εκτός ισορροπίας. Δεν υπάρχουν άλλες υποψηφιότητες, οπότε επίσημα σας ζητώ να ψηφίσετε για τη θέση πέμπτου αντιπροέδρου. Μόνο μία υποψηφιότητα έχουμε. Διαβοής λοιπόν. Ψηφίζουμε αυτή την υποψήφια. Σας ευχαριστώ. Μπορείτε να πάρετε φωτογραφία του Προεδρίου που σχηματίστηκε. Και μετά θα τα ξαναπούμε για πρώτη επίσημη συνειδήση της Επιτροπής στις 22 Ιουλίου. Στο Πανίδιν θα τα πούμε τότε.